και η διαδικασία των ψηφοφοριών. Ο κύριος Αϊκάουτ ε, θα πρέπει να σταματήσετε τις συζητήσεις με τους συναδέλφους γιατί είναι η σειρά που να μιλήσετε. Α, όχι, όχι, βεβαίως. Ξεκινάμε κατευθείαν. Έχουμε λοιπόν την έκθεση Αϊκάουτ. Μέχρι να πέσουν οι τίτλοι, νομίζω ότι θα ηρεμήσουν και οι συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά... Α, ναι, δεν έχει έρθει όμως η Επιτροπή. Να περιμένουμε λοιπόν. Así, donc. Euh, Συνάδελφοι, ας προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Παρακαλώ πολύ όσοι συζητούν στους διαδρόμους ε, ή να διακόψουν ή να συνεχίσουν αλλού. Επίσης οι κλητήρες παρακαλώ να κάνουν αυτή τη δυσάρεστη δουλειά που έχουν που είναι όμως πολύ χρήσιμη. Euh, euh, κύριε Άικχαουτ, θα σας δώσω το λόγο. Μια και είναι η σειρά της δικής σας έκθεσης. έκθεση. Ε, πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές διοξιδίου του άθρακα των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Για τέσσερα λεπτά έχετε το λόγο, κύριε Άικχαουτ. Thank you for all the interest. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ενδιαφέρον που δείχνετε για το διοξιδίτη του άνθρακα και τα φορτηγά, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλά κάνετε και το προσέχετε το θέμα αυτό, γιατί είναι η τελική νομοθεσία την οποία καλούμε να εγκρίνουμε στην τρέχουσα θητεία. Αυτό τι σημαίνει ότι πέρα από την νομοθεσία αυτή θα κληθούμε να κάνουμε πολλέ βελτιώσει, αλλά εδώ χρειάζεται να γιορτάσουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ρυθμίσει τι του άνθρακα, τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Όπω έγινε και με τα ΙΟΤΑΧΗ, ήταν ε, δύσκολο ο αγώνα, μεγάλη αντίσταση που αντιμετωπίσαμε. Καταφέραμε, θεωρώ όμω, με καλή συνεργασία με του διάφορου κοιόδε συζητητέ από τι πολιτικέ ομάδε να ευχαριστήσω για τη συμβολή σα και τη συνεισφορά σα. Δεν συμφωνούσαμε πάντα αλλά νομίζω ότι σε τελική ανάλυση πετύχαμε μια συμφωνία την οποία όλοι υποστηρίζουμε. Και έχουμε την αίσθηση ότι πραγματικά αγγίζουμε το σημαντικό πυρήνα του θέματος αυτού. Και βλέπουμε λοιπόν μείωση του διοξιδίου του άνθρακα 25% μέχρι το 2025. Μέχρι το 2030 δεσμευτικό στόχο 30%. Και ιδιαίτερα αυτή η μακροπρόθεσμη προοπτική θα δώσει ένα σαφές μήνυμα προς τους αυτοκινητοπαραγωγούς, παραγωγούς ε, βαρέων οχημάτων, ότι θα χρειαστεί να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες. Επίσης, καταφέραμε να κλείσουμε και όλα τα παραθυράκια σε ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά τις υπερπιστώσεις αυτές, ε, σε ό,τι αφορά τα υπερπιστωτικά όρια. Και έτσι λοιπόν ε, σε ό,τι αφορά τι τεχνολογίε καύση, σε ό,τι αφορά την επένδυση σε νέε τεχνολογίε για το μέλλον. Το μέλλον το οποίο μπορεί να αποτελεί και υδρογόνο αλλά και άλλε μορφέ ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι μια σαφή ε, καθοδήγηση προ του παραγωγού. Ήταν σκληρό ο αγώνα και προφανώ από πλευρά των πρασίνων θα θέλαμε να έχουμε πιο φιλοδοξού στόχου επιτάπητο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει σαφήνεια μακροπρόθεσμη πλέον για του παραγωγού, προκειμένου να ξέρουν πού οδεύουν και πού θα πρέπει να επενδύσουν. Για να εξασφαλίσουν και ότι το μέσο των μεταφορών επίση καθαρίζει και κινείται προ την ε, μείωση της χρήσης του άνθρακα, γιατί όταν ρωτάμε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο κλάδος, να σας πω ότι είναι 6% του συνολικού ε, των συνολικών επενδύσεων, αλλά σε σχέση με τις οδικές μεταφορές μιλάμε για 25% ποσοστό. Μιλάμε λοιπόν για μια πολύ σημαντική κατηγορία η οποία επιπλέον αυξάνεται η σημασία της. Μέχρι το 2050 ξέρουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μειώσει και να έχουμε αφαιρέσει τον ανθρακά από την οικονομία μας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτή η νομοθεσία. Θα γίνουν αναθεωρήσεις μέχρι το 2022. Να σας ε, υποσχεθώ ότι μέχρι τότε θα κοιτάξουμε και τους στόχους που θα, έχουμε, θα θέσουμε αύριο και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να κάνουμε και πολύ παραπάνω. Γιατί θα δώσουμε ένα σαφές μήνυμα, όπως σας είπα αύριο. Και αλλάζει λοιπόν η αγορά. Έχουμε νέε θέσει οι οποίε θα προκύψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πραγματικά ήταν η σωστή στιγμή να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπω ε, άλλε χώρε, ε, μάλλον όπω η Ιαπωνία, η ΙΠΑ, ο Καναδά έχουν ήδη ρυθμίσει το θέμα αυτό Ουσιαστικά λοιπόν τώρα προσπαθούμε να προλάβουμε αυτές τις χώρες αυτές. Χρειαζόμαστε λοιπόν την κατάργηση του άνθρακα στον τομέα του μεταφορών αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Είναι λοιπόν καλή η έκθεση. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, την Επιτροπή, το Συμβούλιο που απουσιάζει για τη στενή συνεργασία και προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η Και τώρα το λόγο έχει ο έπιτροπο, ο κ. Κανιέτα. Madam President, honorable members. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα για την τελευταία συζήτηση για αυτό το νομοθέτημα. Η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικό επιτεύγμα και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός ε, φιλόδοξου ε, πλαισίου για την ε, καθαρή ενέργεια για το 2030. Αυτή η συμφωνία κατέστη δυνατή χάρη στις προσπάθειες, επικοδομητικές προσπάθειες και των δύο οργάνων. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή τον κύριο Έικχαρτ και όλους τους συνεισηγητές για αυτή την επιτυχία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η συμφωνία η οποία επετεύχθη είναι ισορροπημένη και φιλόδοξη. Τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι ότι για τα νέα βαρύ επαγγελματικά οχήματα η, ο μέσος όρος των εκπομπών το 2025 θα είναι 50% χαμηλότερος σε σχέση με τις, αυτές του 2019. Τα βαρέα οχήματα αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών εκπομπών των επαγγελματικών οχημάτων και ε, ξεκινώντας από το 2019 με τα υπερπιστωτικά μόρια ε, θα μειώσουμε στο 0 τις ε, εκπομπές. Το 2022 θα γίνει μια συνολική επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας αυτής. Αυτό το κείμενο συμπληρώνει την εικόνα. Ο τομέας των οδικών μεταφορών κινείται σαφώς προς, προς μια πιο καθαρή λειτουργία. Τα βασικά ωφέλη είναι ότι οι εκπομπέ βαρέων οχημάτων θα αντιπροσωπεύουν το 25% ε, των συνολικών οδικών μεταφορών. Ε, αυτή τη στιγμή θα αυξηθούν κατά 10% το 2030 αν δεν κάνουμε τίποτα. Με τους στόχους μας όμως και με τους ε, μας στόχους θα μειωθούν κατά 24% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2005. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τους ε, συνολικούς στόχους που έχουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις του Παρισιού. Επίσης θα γίνουν εξοικονομήσεις ε, από πλευράς των ε, ιδιοκτητών τους. Ε, Ξενομήσεις λόγω φθηνότερου καυσίμου. 6.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μεταφορών ε, που δίνουν δουλειά σε 2 εκατομμύρια άτομα θα βοηθούν πάρα πολύ. Επίσης η αυτοκινητοβιομηχανία θα ενισχύσει την καινοτομία της και τη, θα διοχετεύσει καλύτερα τις επενδύσεις της. Δίνουμε κίνητρα για, μηδενικό, για οχήματα μηδενικών εκπομπών ε, ενώ δίνουμε το μήνυμα ε, ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, υποδομές επαναφόρτισης. Τέλος, θα αυξηθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη και θα μειωθούν οι εισαγωγέ πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας καλέσω να στηρίξετε αυτή την συμφωνία αύριο. Θα βάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση προ την κατεύθυνση της μετάβαση προς τις καθαρές μεταφορές. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η Κομισιόν έχει υποβάλει και δύο δηλώσει που ε, προκειμένου να στηρίξει τη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και ε, Κοινοβουλίου. Ε, θέλω να ευχαριστήσω μία ακόμα φορά όλα τα μέλη για τη στήριξή τους. Ευχαριστώ. Κυρία Βίρκουνεν, εκ μέρους Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματο τη Επιτροπή Μεταφορών και να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για το καλό παράδειγμα, ε, συγγνώμη, για το καλό αποτέλεσμα που πετύχαμε. Από πλευρά τη Επιτροπή ε, Μεταφορών ε, έχουμε να πούμε ότι και η παραγωγή ε, βαρέων οχημάτων θα πρέπει να φροντίσουν για μείωση 25% μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030. Είναι φιλόδοξο ο στόχο, αλλά πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκδίδουμε τέτοιε προδιαγραφέ εκπομπών για τέτοια φορτηγά. Και φυσικά, ω τώρα υπήρχαν κίνητρα για την ε, αποτελεσματικότητα και την αποβατικότητα των οχημάτων και για το κόστος, τη μείωση του κόστους ε, των καυσίμων των φορτηγών. Αλλά με τις διατάξεις αυτές θα προσθεθούν περαιτέρω και οι καινοτομίε στον τομέα αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρξουν και μέθοδοι μέτρησης όλες ε, Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη η κατανάλωση ενέργειας σε όλο τον ε, κύκλο παραγωγής, γιατί έχουμε μεγάλο περιθώριο μείωση των εκπομπών στις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στις πολιτικές ομάδες. Έχουμε τον κύριο Φιέλνερ από το ΕΛΚΑ. Για δύο λεπτά ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σε... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ολοκληρώνονται πολλά χρόνια δουλειά και για μένα και για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο. Αύριο θα εγκρίνουμε τους κανόνες. Ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά το αποτέλεσμα είναι θετικό. Έχουμε καλύτερες μεταφορές χωρίς μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αυτή είναι η τελευταία φορά που απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για 15 πανέμορφα και εξαιρετικά χρόνια. Άρχισα να γκριζάρω νεκρό ταφί μου όλα αυτά τα χρόνια εδώ και άλλοι και άλλων, αλλά ήταν τιμή μου να εκπροσωπώ τη Σουηδία και το κόμμα των συντηρητικών μπορέσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς όφελος του ελεύθερου εμπορίου που βγάζει τους ανθρώπους από τη φτώχεια, κάνει πλουσιότερη την Ευρώπη, να βελτιώσουμε το περιβάλλον, τον, φέραμε τον άνθρωπο στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων, αλλάξαμε την Σουηδία, αλλάξαμε τα πράγματα και για την Ευρώπη. Μπορεί να μην ήμουν πάντα ένας μετριοπαθής, αλλά πάντα προσπάθησα να προασπίσω την το σωστό και τους ψηφοφόρους μου. Γιατί πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι κάτι που αξίζει να πολεμήσουμε για την ειρήνη και την κοινότητα. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι αυτή είναι η βασική ελπίδα για την οποία πρέπει να δουλέψουμε. Ευχαριστώ. La parole est à Monsieur δύο λεπτά για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Καλύτερα με το μικρόφωνο, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει μικρόφωνο, κύριε Τζόφολη. Συνεχίζετε να μην έχετε μικρόφωνο. Με ακούτε τώρα. Η ο κανονισμός που υποστηρίζουμε παρά τα προβλήματα που έχει ε, ε, ε, φέρνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά από πολλές αντιστάσεις κοινά όρια για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρωπου για τα βαριά επαγγελματικά οχήματα που συμβάλλουν κατά 6% στις συνολικές εκπομπές της Ένωσης, εκπομπές που προβλέπεται να αυξηθούν. Πέρα των target στόχων που είναι φιλόδοξοι αλλά μπορούμε να, τους πετύχουμε, έχουμε μια σειρά πρότυπων επιδόσεων στο δρόμο με εκπομπές για την κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Αυτά τα πραγματικά στοιχεία συχνά απομακρύνονται από αυτά που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και είναι αναγκαία για να αποφύγουμε στρεβλή συμπεριφορά και τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τρίτους για ελέγχους, για ανεξάρτητους ελέγχους. Κατά Σημαντικό είναι το αίτημα της Επιτροπής μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της, της, ε, ε, των εκπομπών των οχημάτων αυτών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωή τους. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ένα μηχανισμό κινήτρων για την διάδοση ηλεκτρονικών φορτηγών ή χαμηλής, χαμηλών εκπομπών για να εξασφαλίσουμε από το 2025 ένα υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό των οχημάτων αυτών ε, στο ύψος του 2%. Θα δοθούν κίνητρα σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και υποδομές για, την ηλεκτρική, για τα ηλεκτρικά φορτηγά στην πορεία για την ε, απομάκρυνση από τον άνθρακα που κατά 94% εξαρτάται ακόμα και τώρα από το πετρόλαιο θα πρέπει να εξετάσουμε και το ρόλο του φυσικού αερίου. Είναι αναγκαίο ωστόσο η Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ταμείο για την πανακατάτηση ε, ε, των εργαζομένων στον κλάδο για να καταστήσουν την βιώσιμη, τη μετάβαση βιώσιμη και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Ο αυτός αποτελεί ένα επιπλέον βήμα σε μια Ευρώπη που αλλάζει προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στη συμμαχία μεταξύ βιομηχανίας και περιβάλλοντος. Ο κ. Μάκρη, για 1,5 λεπτό. Αύριο το μεσημέρι έχουμε την τελευταία ε, ψηφοφορία της τρέχουσας και πάλι έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε για συγκεκριμένα μέτρα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τα φορτηγά είναι ευθύνονται για 6% των συνολικών εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ένα τέταρτο των ε, οδικών μεταφορών. Και αυτές οι εκπομπές αυξάνονται ακόμα και στη δική μου χώρα, στη Φλάνδρα. Θέλουμε, αν θέλουμε λοιπόν ε, να πετύχουμε τους στόχους μας και τις δεσμεύσεις μας για το κλίμα, θα πρέπει να πρασινίσουμε τον στόλο μας. Έχουμε την τεχνολογία αυτή. Είναι κρίσιμη σημασία, καταρχάς, να υπάρξει ένα πρότυπο μείωση του διεξιδίου άνθρακα για τα φορτηγά και τα κίνητρα για να ενθαρρυνθούν τα φορτηγά χαμηλών εκπομπών. Είναι σημαντικό και γι' αυτό λοιπόν το κόμμα μου το ΕΝΒΑ υποστηρίζει αυτή την τελική νομοθεσία παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε πιο υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας. Το πρασίνισμα λοιπόν του στόλου είναι πολύ σημαντικό για καλύτερη ποιότητα της ατμόσφαιρας γιατί αυτή προκαλεί θανάτους πρόωρους. Τα πρότυπα αυτά φροντίζουν να υπάρχει και μείωση ε, του κόστου των καυσίμων. Αυτό είναι καλό για το καταναλωτή. Και τέλος, ε, η φιλόδοξη αυτή θέση προτύπων ε, χρειάζεται για να προσελκύσουμε επενδύσεις και κοινοτομία. γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ο κύριος Τόρβαλτς για δύο λεπτά έχει το λόγο από την Άλτα. Πρόεδρε, ξεκινώ ευχαριστώντας τους συντρόφους και συναδέλφους που δούλεψαν μαζί μου αυτά τα χρόνια στις διαπραγματεύσεις. Είχα συνεργαστεί με τον κύριο Άικχαουτ και τον Κρίστο Φιέλνερ. Γκρίζαν τα μαλλιά του, είπε ο κύριος Φιέλνερ, αλλά αν δω τον Επίτροπο ή και εμένα στον καθρέφτη θα έλεγα πολύ περισσότερα γκρίζα μαλλιά έχουν άλλοι. Έχουμε μπροστά μας κάποιες σημαντικές προκλήσεις. Πρώτον, κατακαιρματισμός στην κατασκευαστική διάσταση. Πολλοί κατασκευαστές θα τηρήσουν τους στόχους χωρίς δυσκολία, άλλοι θα το πετύχουν πολύ πιο δύσκολα και θα δυσκολεύσουν έτσι τα πράγματα. Άλλο πρόβλημα είναι τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, όπως τα λέμε. Το, τα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών, αλλά με βρώμικο ηλεκτρισμό, δεν είναι και πολύ καθαρά. Πρέπει να έχουμε λοιπόν σημαντικούς στόχους, ε, όπως αυτούς που συζητήσαμε χτες με την Κρέτα Τούμπεργκ αν θέλουμε θα πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι ο δρόμος μπροστά. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια γέφυρα για το μέλλον με εναλλακτικά καύσιμα, εξασφαλίζοντα ότι οι εκπομπές, ε, τα όρια των εκπομπών είναι χαμηλότερα από αυτά του ηλεκτρισμού που χρησιμοποιούμε σήμερα. Η μεγαλύτερη πρόκληση προ τα εμπρό έχει να κάνει με αυτό που είπε στο ξεκίνημα τη παρέμβαση του ΟΜΠΑΣ, την παρακολούθηση τη εφαρμογή τη νομοθεσία αυτή τα επόμενα έτη. Μιλάμε τώρα για το επόμενο κοινοβούλιο, το οποίο θα έχει έτοιμη δουλειά εξασφαλίζοντας ότι η πρόταση αυτή θα φτάσει στην, τον προορισμό που έχει και ότι η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι θα γίνονται τα σωστά πράγματα. Ο Μπάς και άλλοι που μπορεί να είναι εδώ θα μπορέσουμε αν θέλουμε να βοηθήσουμε την υλοποίηση αυτής της, ε, ε αυτής της Κάποιο ε, ζητάνε να δέξει να απαντήσετε μια μπλε κάρτα. Πάντα με χαρά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συναδελφό, τον κύριο Τόρβαλτσε, γιατί το διοξείδιο του ανθρακά προφανώς και αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Και γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να δούμε και το κύκλο, σε όλο τον ε, κύκλο παραγωγής των φορτηγών. Και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και τι γίνεται με τα χρησιμοποιημένα φορτηγά. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα διαρκές ε, τέτοιο ζήτημα στις ε, πόλεις και αυτά θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σημείο το οποίο χρειάζεται ο δεν είναι τόσο τα ευφύ οχήματα, αλλά κυρίως οι ευφύς οδηγή. Δεν ξέρω που μπορεί να βρει φυσικά ο κύριος έχει ευφύ οδηγούς. Αλλά αυτό χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να μας ε, εκπαιδεύσουν στην οδήγηση. Χρειαζόμαστε τεχνικά εργαλεία για να έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο και να μην φοβούμαστε την τεχνολογία και όλε τις ευκαιρίες που παρέχει. Αν δεν φοβόμαστε, θεωρώ ότι μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, ο κύριος Εκ. 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Συχνά άσκησα κριτική στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά ε, τις αποφάσεις προς όφελος των μεγάλων ομίλων και προς ε, εις βάρος ε, της, του ανθρώπου, των, των ζώων και του περιβάλλοντος. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που πέτυχε ο εισηγητής, ο κύριος Αικχάουτ. Αύριο θα ψηφίσουμε για τον πρώτο κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα φορτηγά. Παρά της μεγάλης αντίδρασης της, του οικονομικού κλάδου και πολλών κυβερνήσεων και κυρίω τη γερμανική κυβέρνηση, αυτή η πρόταση ξεπερνά κατά πολύ την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντο. Δεν επαρκεί, ασφαλώ. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά να κάνουμε σε πολλού τομεί. Σήμερα είναι η τελευταία μου ομιλία αυτή εδώ στην Ολομέλεια. Δεν πρόκειται να είμαι βουλευτή στην επόμενη θετία. Θα σα καλέσω λοιπόν να τηρήσουμε το άρθρο 13 της Συνθήκης Λισαβόνας και να λάβουμε υπόψη την ευημερία των ε, δισεκατομμυρίων ζώων, τα οποία τη χάνουν εκμετάλλευση και ε, τα θανατώνουμε, να κάνετε πολιτική με την καρδιά σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσετε φυσικά και το κουμπί της λογικής θα πρέπει να αλλάξουν τα πολιτικά παράδειγματα. Να μην κοιτάμε μόνο την οικονομική ανάπτυξη, να μην είναι μόνο αυτό απότερο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ευημερία, η ευτυχία όλων των ε, ζώων, των οργανισμών και των ζώων. Αυτό αναμένουν οι πολίτε από εσά. Αυτό προσδοκούν οι πολίτε από εσά. Σα ευχαριστώ. Να είστε καλά και να έχετε το χέρι στην καρδιά στι μελλοντικέ πολιτικέ αποφάσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμη κυρία συναδελφέ, κυρία Έξα, Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα για το μέλλον προσωπικά. Έχω μία ερώτηση όμως να σας κάνω παρόλα αυτά. Αυτές τις πληροφορίες, από πού τις έχετε πάρει ότι αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας ξεπερνούν κατά πολύ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό ζήτησε και η γερμανική κυβέρνηση 15% και 30%. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχος ο στόχος και δεν ξεπερνά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξή ότι σε κάποια σημεία στις διαπραγματεύσει πετύχαμε στόχους οι οποίοι ξεπερνούν ε, σίγουρα κατά πολύ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό το οφείλουμε κυρίως στον πολύ καλό συνάδελφό μα, τον εξαιρετικό συνάδελφό μα τον κύριο Έκα, ο οποίο πολέμησε με νύχια και με δόντια προκειμένου να είναι φιλόδοξη η έκθεση και γι' αυτό θα ήθελα προσωπικά να του απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, Ντέλη. Η κυρία Ντέλη έχει το λόγο. Παρακαλώ, Καρύμα. Συνάδελφοι, αυτή την εβδομάδα δεχθήκαμε στο Κοινοβουλίο την Κρέτα Τούμπεργκ που ήρθε να μας πει αναλάβετε δράση, κάντε κάτι, κάντε κάτι τώρα. Φροντίστε ότι εσείς που αποφασίζετε να επιτρέψετε να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να ζήσουν ευτυχισμένες σε έναν φιλόξενο κόσμο. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τον πλανήτη και την υγεία μας, θα πρέπει να, και να μειώσουμε την ρήπανση, θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και να υποχρεώσουμε τον κλάδο των μεταφορών να συμβάλλει όπως οι άλλοι. Στους δρόμους της Ευρώπης 5% ε, είναι μόνο τα φορτηγά μεταξύ των οχημάτων που παράγουν ωστόσο το 27% το 1 τέταρτο δηλαδή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα των οδικών μεταφορών στην Ένωση. Αν θέλουμε μια μέρα να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις του COP21 να σώσουμε, για να σώσουμε το κλίμα και τον πλανήτη είναι καιρός να σταματήσουμε με αυτή την ανισορροπία. Με το κείμενο που υποβάλλεται ψηφίζουμε και κάνουμε τα πρώτα βήματα για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, λιγότερα ε, ε, αέρια μέχρι το 2000, με μείον 15% για τα φορτηγά. Ο κανονισμός πάει παραπέρα από την πρόταση επιτροπή και για πρώτη φορά δεσμεύει την Ευρώπη να μειώσει την ε, ρήπανση των μεγάλων φορτηγών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι νικήσαμε. Τι δείχνει αυτή η νίκη. Δείχνει ότι όταν εμείς οι ψηφοφόροι Ακούμε τα αιτήματα, ιδίω τη νεολαία που κάθε εβδομάδα κάνει απεργία για να σώσει το κλίμα. Όταν εγκρίνουμε ε, όταν περνάμε από τα ωραία λόγια σε συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, προσοχή ωστόσο. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την δυνατότητα τα παιδιά μας να ανασάνουν, να ζήσουν ελεύθερα, να χαρούν αυτό τον ωραίο πλανήτη, θα πρέπει αύριο να ψηφίσουμε το κείμενο αυτό, γιατί ψηφίζοντας το κείμενο ψηφίζουμε για το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για την Ευρώπη των Εθνών και Ελευθεριών. Λαντσίνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κλάδος της κίνησης είναι θεμελιώδης και για την οικονομία και για την κοινωνία των κρατών μελών. Ωστόσο εδώ συνεχώς ξεχνάμε αυτή τη διάσταση και δεν ακούμε τα αιτήματα των επιχειρηματιών και εργαζομένων. Τα μέτρα που περιλαμβάνει η πρόταση αυτή είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων αναχρονιστικά ή, ή ε, παράλογα. Μιλάμε για μια βιώσιμη μετακίνηση προς την κινητικότητα χωρίς κατανάλωση, χωρίς όμως να κάνει μια αξιολόγηση των αντικτύπων των μέτρων που προτείνονται. Το μέτρο μιλά, υποχρεώνει να στραφούμε στα ηλεκτρικά, εξαφανίζοντας και αγνώντας τις άλλες εναλλακτικέ λύσεις που υπάρχουν στην αγορά. Θα έπρεπε εξ αρχής να προβλέπεται η χρήση μείγματος τεχνολογιών και μεγαλύτερες προθεσμίες για να διευκολυθούν οι επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών εκπομπών ε, μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα, ιδίω ό,τι αφορά τα ε, μεγάλα τα φωτιγά. Ο κλάδος θα πληγεί εις βάρος της ευρωπαϊκής ε, και των κρατών μελών. Η Ευρώπη θα γίνεται ακόμα περισσότερο ε, εξαρτημένη από τρίτες χώρες για την απακτήση ε, μπαταριών. Και Επιπλέον, όπως αναφέρει ο τύπος και παράδοξα, χρησιμοποιήθηκαν μόνο ε, νέες στήλε για ε, ηλεκτρική ενέργεια που όμως τροφοδοτούνται από δίζελ. Ε, ο κλάδος της, της, της οδικής κίνησης θα μπορούσε να χάσει ε, μόνο στη Γερμανία μεταξύ 75.000 και 210.000 ε, μονάδων μέσα στο 2030. Σκεφτούμε καλύτερα την πρόταση αυτή που όπως διατυπώνεται αυτή τη στιγμή στην ουσία είναι ακατανόητη και με αποτελέσματα αντίθετα από αυτά που έχει θέσει ως στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σόσνιετς. Ένα λεπτό. Ε, στα έγγραφα μιλάμε συνεχώς για μηδενικές εκπομπές, αλλά μηδενικές εκπομπές δεν υπάρχουν ούτε θα υπάρξουν. Είναι ένα εργαλείο marketing που χρησιμοποιείτε εσείς ή αυτοκινητοβιομηχανίες. Μεταφορές μηδενικών εκπομπών δεν είναι δυνατές. Κάποιο ε, ε, κάποιος θα εκπέμπει. Αν δεν εκπέμπουν τα οχήματα θα εκπέμπουν οι βιομηχανίες οι οποίες θα παράγουν την ενέργεια που χρησιμοποιούν τα οχήματα. Οπότε πολύ ωραία να δράσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή η τεχνολογία δεν μας επιτρέπει να φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές. Κάπου θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και θα χρειαστεί να μεταφερθεί. Μηδενικές εκπομπές δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν η έκθεση αυτή είναι ανεύθυνη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λίζα. Ενάμιση λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Και είναι πολύ καλό το γεγονό ότι αύριο για πρώτη φορά ορίζουμε όρια για τι εκπομπέ των βαρέων οχημάτων. Γιατί όλοι τα θα πρέπει να συμβάλλουν αυτό που του αναλογεί στη μείωση των εκπομπών. Είναι φιλόδοξο αλλά εφικτό το σχέδιο που έχουμε μπροστά μα και είναι καλό που έχουμε που δεν υποκύψαμε στις υπερβολικές ε, ε, απαιτήσει των πράσινων στο κείμενο αυτό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μπάς για την ε, ρεαλισμό που έδωσε, γιατί ήθελε πολλά παραπάνω αρχικά, αλλά επικεντρώθηκε στα ουσιαστικά και αυτό ήθελε και το ΕΛΚ, αυτό ήθελε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν ευφυέ αυτό. Να ευχαριστώ και τον κ. Φιέρνερ για την δέσμευσή του, όχι μόνο για το θέμα αυτό, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Αλλά θα ήθελα να πράξω την ευκαιρία όλος ιδιαίτερος για να ευχαριστήσω και τον Επιτρόπο κύριο Κανιέται, γιατί στην ακρόαση, ακρόαση του αντιμετώπισε τα πειρά της κριτικής και τότε ακόμα και αυτοί που τον επέκριναν τότε θα πρέπει σήμερα να ομολογήσουν ότι πετύχαμε πολλά μαζί για την προστασία του κλίματος στην Ευρώπη και είναι η τελευταία νομοθεσία που θα περάσει το Κοινοβούλιο αυτό. Γι' αυτό να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον Επιτροπό, τον κύριο Κανιέτε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και ένα θέμα νομίζω που θα χαρακτηρίσει την επόμενη περίοδο είναι η ενίσχυση των συντροδρόμων. Καλό είναι να ρυθμίσουμε και τα φορτηγά, αλλά θα πρέπει όλο και πιο πολλά εμπορεύματα και ε, επιβάτες να μεταφερθούν στο συντροδρόμο και να δούμε ότι σε ό,τι αφορά την ε, μείωση των εκπομπών είναι πολύ πιο επιβαρημένος ο συντροδρόμος από ότι οι άλλοι τομεί μεταφορών. Και εδώ θα πρέπει κάτι να κάνουμε λοιπόν στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Και κύριε Λίζα, έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Σόσνη, έτσι. Την αποδέχεστε βεβαίω. Με χαρά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Πολλά πατήχαμε. Πετύχαμε σε ό,τι αφορά το κλίμα σε ό,τι αφορά κάποια στερεότυπα τα οποία πέρασαν στο κλίμα. Τι θα σημαίνουν όμως όλα αυτά συγκεκριμένα για το κλίμα, ο κύριος Λίζε. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά όταν ε, μου κάνετε την ερώτηση αυτή να σας το πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει τις στόχους της για το 2030 και αποφασίσαμε λοιπόν για μια νομοθεσία και αύριο θα αποφασίσουμε το τελευταίο τμήμα της νομοθεσίας αυτής, όπου ο νομοθετικός πώς δημιουργούμε τους όρους για να εκπληρώσουμε και με το παραπάνω τους στόχους μας για το 2040. Είναι απαραίτητο λοιπόν η Ευρώπη να αποτελέσει πρότυπο και για τις άλλες επίρρους και παράλληλα έχουμε και κανόνες που δεν θα διώξουν τη βιομηχανία από την Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό είναι καλή ισορροπία και όταν έχουμε τα βέλη τη κριτική και από τι δύο πλευρέ του πολιτικού φάσματο, αυτό είναι καλό δείγμα ότι είναι ισορροπημένη η νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντάλη για 1,5 λεπτό. Μυρία, μου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον εισηγητή μα, τον κύριο Άικχαουτ, για τη δουλειά που έκανε και το συμβιβασμό που πέτυχε, γιατί ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο ο φάκελο αυτό. Ήταν πάρα πολύ το γεγονό ότι έχουμε πλέον άλλη μία πολιτική για τη μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όπου δεν είχαμε πρότυπα για τα ε, βαρέα οχήματα. Παρά το γεγονό ότι γνωρίζαμε την μεγάλη επίπτωση που έχουν τα φορτηγά αυτά στην ε, παγκόσμια αύξηση του θερμοκρασία. Και αυτή αναμένεται να αυξηθεί. Έχει έρθει λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να εγκρίνει δεσμευτικά πρότυπα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών. Ήταν λοιπόν δύσκολο το έργο αυτό. Η διαπραγμάτευση για το Συμβούλιο, με το Συμβούλιο για την θέση των benchmarks ήταν πραγματικά μεγάλο επιτεύγμα. Το ξέρω αυτό από προσωπική εμπειρία να ευχαριστήσω και τον εισηγητή από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τον κύριο Τσόφολη, για την μεγάλη του δέσμευση και τον ρόλο που έπαιξε για να πετύχουμε συμβιβασμό. Η θέση του Κοινοβουλίου θέτει το σωστό επίπεδο φιλοδοξίας. Αυτό χρειάζεται για να ε, καταφέρουμε να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας για το κλίμα και πιστεύω ότι το μέλλον των καθαρών οχημάτων και των φορτηγών θα καθοριστεί από την κοινοτομία μόνο με ισχυρά κίνητρα για την παραγωγή οχημάτων χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών τελικά θα περάσει την αλλαγή αυτή. Αυτό αποτελεί το σκόπο μας και το στόχο μας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με τη δουλειά μας και προσβλέπω και τις μελλοντικέ μας προσπάθειες τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο λόγος στην συνάδελφο εγώ Νταλόντα για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε. Επιτέλους ε, καθορίζονται ε, στόχοι μείωσης ε, εκπομπών για τα, βόρεια, για τα βαριά οχήματα. Ε, Τέτοιου είδου στόχου και πολύ πιο φιλόδοξου είχαμε στηρίξει εμεί στην Επιτροπή Μεταφορών. Όμω η Γερμανία και άλλε χώρε πιεσμένες από την αυτοκινητοβιομηχανία τους μείωσαν τους ε, στόχους. Παρ' όλα αυτά, οι εκπομπέ διοξείδου του άνθρακα συνεχώ αυξάνονται τα τελευταία χρόνια στι οδικέ μεταφορέ. Αντίθετο, η αναθεώρηση του 2022 θα είναι πάρα πολύ σημαντική, προκειμένου να προσαρμόσουμε την νομοθεσία και ενδεχομένω να καλύψουμε περισσότερου τύπου οχημάτων και ενδεχομένω να ξαναδούμε ε, του στόχου μα. Παρόλο υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης από τα κράτη-μέλη. Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα οδικό χάρτη υποχρεωτικό. Ο κανονισμός αυτός είναι ένα βήμα για να καταπολεμήσουμε την ατμοσφαιρική μόλυνση και να σεβαστούμε τους κλιματικούς στόχους, ιδιαίτερα του Παρισιού, που θα περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Αυτό προς όφελος των επόμενων γενιών. Η Ευρώπη δρά με συγκεκριμένο τρόπο κατά της μόλυνσης και τελευταία μου αυτή ομιλία στην Ολομέλεια θέλω, θέλω να υπογραμμίσει ακριβώς αυτή την πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κάτσε διάει. Δύο αιτήματα έχουν ε, γίνει δεκτές, έχουν υποβληθεί. Φάρια. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Εκχάουτ και όλους τους συναδέλφους ε, που βοήθησαν να θέσουμε τέτοιους φιλόδοξους στόχους για τα βαρέα οχήματα. Επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας για διαφορετικά χαρτοφυλάκια, διαφορετικούς φακέλους ε, που έχουν σχέση με τους στόχους του Παρισιού, την κυρία Ντάλη πιο συγκεκριμένα. Είχαμε κάνει πρόταση για πιο φιλόδοξους στόχους και ελπίζουμε ότι αυτές οι προτάσεις, ε, οι προτάσεις του ΕΛΚ ε, βοήθησαν. Προφανώς η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Πρέπει να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας και να μειώσουμε την τοξικότητα της ανθρώπινης δράσης στον πίνακα. Οι επιστήμονες ε, στέλνουν σήμα κινδύνου στην κοινωνία αλλά ε, υπάρχει κάτι το οποίο κάνουμε, ε, δεν κάνουμε σωστά. Δεν προχωράει αρκετά γρήγορα η μείωση της χρήσης του ε, άνθρακα. Κέλλη, e το λόγο. Ασχολούμαι με θέματα κλιματικά καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας. Και χαίρομαι για την πρόοδο που κάναμε στο Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια στον Επίτροπο Κανιέτε. Και τον κύριο Αικχάουτ που αποτέλεσε ατμό μηχανή σε αυτό το τομέα τα τελευταία πέντε χρόνια. Όπως είπε η Μύρια Μτάλη, ε, έχουμε πλέον μια πολιτική για τα βαρέα οχήματα. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές. Όσο βελτιώνεται η οικονομία, ε, εγώ πηγαίνω από το, από το, το σπίτι μου στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου και από το Στρασβούργο στη Φραγκφούρτη και βλέπω όλο και περισσότερα βαρύ οχήματα στους δρόμους. Η μείωση αυτή που προβλέπουμε δεν σημαίνει ότι θα, θα μειωθούν οι μεταφορές. Απλά θα τις κάνει πιο α, ενεργειακά αποδοτικές. Οπότε μπορούμε να γίνουμε πιο φιλόδοξοι τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι μια καλή αρχή. Είναι μια λογική πρόοδος, προοδευτική, σταδιακή και νομίζω με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουν το περιβάλλον μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Thank you very much. Ολοκληρώνει τη διαδικασία του Κατσδιάη. Το λόγο τώρα για την Επιτροπή ο Επίτροπος Άριας Κανιέται. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές για τη συζήτηση αυτή. Να απαντήσω σε μια απευθεία ερώτηση που μου έφεσε ο κ. Σόσνιεκ. Ρώτησε, τι έκανε αυτό το κοινοβούλιο για την αργή του κλίματος. Η απάντηση μου είναι πολλά. Τι έκανε, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αργή του κλίματος. Όχι πολλά. Πριν το 2020 θέσαμε στόχους μείωσης των εκπομπών και το 2017 μειώσαμε τις εκπομπές κατά 17% σε σχέση με το 1990. Μειώσαμε τις εκπομπές, αναπτύξαμε, αναπτύξαμε τα ανανεώσιμα, κάναμε καλύτερη ε, λειτουργία των επιδόσεων, αλλά το κοινοβούλιο αυτό διπλασίασε το πλαίσιο για την ενέργεια. Ήμουν στην πολιτική, είμαι στην πολιτική 38 χρόνια. Έχω έχω, έχω υπηρετήσει σε εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Ποτέ δεν είδα τόσο έντονη νομοθετική διαδικασία ε, διδαστηριότητα όσο εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους των επιτροπών, την κυρία Βάλη, τον κύριο Μπούσεκ, τον Τζοβάνι Λαβία, όλους τους εισηγητές, ξεκινώντας από τον κύριο Άικχαουτ, που έκανε εξαιρετική δουλειά που ήταν και δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις όπως στα ανανεώσιμα. Και αυτό που κάναμε είναι ότι υιοθετήσαμε πολλά νομοθετικά κείμενα που θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών το 2011 κατά 45% και αν αλλάξουν και θα αλλάξουν το 2030 θα έχουν 60% μειώσει των εκπομπών. με μεγάλο πακέτο. Και ένα από τα πιο σημαντικά είναι ο μέσος, το μέσο ποσοστό πολιτικών πολιτική υποστήριξη προτάσει αυτέ. Στο πακέτο ενέργειας 80% των ψηφοφοριών ήταν υπέρ. Στο κλίμα 76%. Σημαντική λοιπόν πολιτική υποστήριξη για την νομοθεσία που υιοθετήσαμε το 2030 που σημαίνει ότι Είχαμε έναν διάλογο, υπήρχε αμοιβαία κατανόηση, υπήρχαν διαπραγματεύσεις και όπως σας είπα ήταν μια απίθανη ευκαιρία. Μετήσχα σε 71 τριμερείς διαλόγους. Δύσκολους που πάνω από 350 ώρες της ζωής μου. Αλλά ήταν εξαιρετικές ευκαιρίες για να μάθω και να σας ευχαριστήσω όλους γιατί η δουλειά αυτή ήταν μια εξαιρετική δουλειά που δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την δική σας εμπλοκή. Εσείς πιέζετε και εμείς ε, απαντάμε. Αυτό είναι ο θεσμικός ρόλος του καθενός. Το βασικό στοιχείο είναι ότι περνάμε ένα κείμενο που θα εφαρμοστεί για την επόμενη 20 ετία, αλλά έχουμε τη δυνατότητα αναθεώρησης καθοδών για με αύξηση των στόχων. Στις 77% των πιθανών ψηφοφόρων για τις ευρωεκλογέ ανέφεραν σε μια σφιγμομέτρηση την περασμένη εβδομάδα ότι το περιβάλλον ήταν ο βασικός λόγος να πάνε να ψηφίσουν τις ευρωεκλογέ. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η αλλαγή του κλίματος είναι ένας βασικός παράγοντας για να συζητηθεί στις ευρωεκλογικέ. Σας παροτρύνω να κάνετε δύο πράγματα. Πρώτον, να εξηγήσετε στους πολίτε της Ευρώπης τι κάναμε αυτά τα πέντε χρόνια. Και επίσης, να πείτε τι θέλετε να κάνετε τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό θα φέρει περισσότερο κόσμο στις κάλπες και θα μπορέσει το Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία να βοηθήσει την ολοκλήρωση του πακέτου, την περαιτέρω πρόοδο και την συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να μπορέσει η Ένωση να γίνει το 2020 η πρώτη μεγάλη οικονομία που θα είναι ε, ε, ενεργειακά ουδέτερη. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα ο κύριος Σάικα, ο εισηγητής. Μπάς, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και καταρχά, μια και βρισκόμαστε σε τέτοια κλίμα ευγνωμοσύνη, να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο, τον Επίτροπο Μαρία Κανιέτα, για τη δουλειά που έκανε. Και προφανώ και είχαμε στιγμέ όπου διαφωνήσαμε και κάποιε από τι ώρε αυτέ τι ε, περάσαμε μαζί. Να πω ότι Ανά πάσα στιγμή ο διάλογο ήταν καλό. Δεν συμφωνούσαμε πάντα, αλλά υπήρχε πάντα αμοιβαίο σεβασμό και αυτό είναι απαραίτητο για το μέλλον. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι πετύχαμε πολλά. Πετύχαμε πολλά για το κλίμα, για την ενέργεια, για την κινητικότητα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει όμω το έργο μα Γι' αυτό, όπω είπατε, δεν έχουμε ακόμα ε, μπει στη σωστή τροχιά για την ε, ε, οικονομία τυφλική προς το κλίμα. Και αυτό θα το τονίσουμε και αύριο. Και είναι ένας από τους λόγους αυτούς για τους οποίους αύριο και στις ευρωεκλογέ. Το θέμα θα είναι το κλίμα, θα είναι οι εκλογές του κλίματος. Και να σας πω, δυστυχώς να δώσω και ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναήλθατε, γιατί μπορώ να σας απαντήσω για το που εμείς ως Κοινοβούλιο κάναμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο φιλόδοξη. Καταρχάς, ο, ο στόχος για το 2030 πλέον είναι νομικά δεσμευτικός. Αυτό δεν ήταν στην αρχική πρόταση. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι σαφές μήνυμα για το που οδεύουμε. Δεύτερον, κλείσαμε πολλά παραθυράκια στις προτάσεις και κυρίως αυτά για τις ε, για τα υπερπιστωτικά μόρια σε ό,τι αφορά τα ε, οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και τρίτων. Ε, σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα για τα οχήματα στον δρόμο, τα βελτιώσαμε για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι αυτά που συμφωνούμε θεωρητικά θα εφαρμοστούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τον Dieselgate. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι τόσο απαραίτητα και τόσο κρίσιμα πέρα από τι τεχνικέ βελτιώσει και τι ρήτρε αναθεώρηση και το καθεξή. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι τόσο σημαντικά λοιπόν που στέλνουν ένα μήνυμα προ του επενδυτέ, του κατασκευαστέ ότι το μέλλον θα είναι μηδενικέ χαμηλές εκπομπές στα οχήματα και ότι αν συνεχίσουν όπως ε, σήμερα δεν θα πάνε μπροστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαστικά λοιπόν καταλαβαίνετε σα έδωσα τι απαντήσει αυτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία να δούμε τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε και μετά. Εν ώψη και τη Συνόδου στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο, γιατί περιμένω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τι ε, εθνικέ τη ε, σύνδρομες βλέπω να προσεύχεται και ο Επίτροπος να ευχηθώ και εγώ για αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Πέρα της συνδρίαση. Και θα γίνει αύριο η ψηφοφορία. L'ordine del giorno reca. Βάσει τη ημερήσια διάταξη, προχωρούμε τώρα στην ε, έκθεση Γκαζίμπ για την πρόθεση καθαρών και ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Δίνω αμέσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Γκαζίμπ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε, κύριε Επίτροπε. Πρόκειται για μια οδηγία που θα στηρίξει τα οχήματα, ε, τα ενεργειακώς πιο αποδοτικά οχήματα. Το 60% ορισμένοι λένε 65-66% της μόλυνσης ε, στις πόλεις λέγεται ότι οφείλεται στον τομέα των μεταφορών. Μπορούμε να βελτιώσουμε τα οχήματά μας, ε, τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά, αλλά υπάρχουν εκπομπές και από αλλού. Και αυτό το βλέπουμε στους, στις κρατικές προμήθειες και στους δημόσιους διαγωνισμούς. Αν εγκρίνουμε αυτό το κείμενο θα εγκρίνουμε πολύ φιλόδοξους στόχους και πρέπει αυτοί οι στόχοι να είναι εφαρμόσιμοι στην πράξη. από τις δημόσιες διοικήσεις. Οπότε είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να στηριχθούν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Οι στόχοι αυτοί λαμβάνουν υπόψη και τις δυνατότητες των διαφορετικών κρατών μελών. Ελπίζουμε να μπορούν να υλοποιηθούν και τα κράτη-μέλη να φτάσουν μέχρι σε αυτό το σημείο. Προφανώς δεν μιλάμε για το 100% των αγορών γιατί υπάρχουν παραδοσιακές τεχνολογίες, σημαντικές τεχνολογίες που δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Οι τοπικέ αρχές μας είπαν, ε, για παράδειγμα, ότι τα υβριδικά οχήματα είναι μια καλή βοήθεια για να μειωθούν οι εκπομπές και να προχωρήσουμε προς μηδενικές εκπομπές. Υπάρχει μια τεχνογνωσία που ήδη είναι γνωστή για αυτά τα οχήματα. Χρειάζεται επίσης να εξασφαλίσουμε μια ελαστικότητα μέσω τη οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα, για παράδειγμα, πρόκειται για κείμενα τα οποία ήδη υπάρχουν. Το κείμενο αυτό αφορά και τα βαρέα και τα ελαφρά οχήματα και θα επηρεάσει και τα λεωφορεία στις δημόσιες μεταφορές. Οι περισσότερες αγορές γίνονται μέσω κρατικών διαγωνισμών, οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία. Η, τα αυτοκίνητα είναι ο βασικός στόχος αυτής της οδηγίας, μπορώ να πω και οι κατασκευαστές των λεωφορείων έχουν πλέον τεχνολογία την οποία θα πρέπει να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο και να την χρησιμοποιήσουν προκειμένου τα νέα λεωφορεία να μπορούν να ανταγωνιστούν στις παγκόσμιες αγορές, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά. Για παράδειγμα, η, ε, η εταιρεία Solaris στην Πολωνία έχει λεωφορεία με μηδενικέ εκπομπές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη αλλά και εκτό Ευρώπης. Ελπίζουμε ότι η τεχνολογία ε, χαμηλών εκπομπών η οποία αναπτύσσεται με τη χρήση βιομεθανίου για παράδειγμα θα επιτρέψει να μειωθούν οι εκπομπές ε, στις ε, δημόσιες μεταφορές. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επωφεληθούμε καλύτερα από το βιοαέριο, τα βιοκάψιμα, κάτι το οποίο θα είναι πολύ θετικό για το περιβάλλον μας. Το βλέπετε αυτό στην πρότασή μου. Στο μέλλον θα κατασκευάζονται οχήματα μηδενικών εκπομπών, αυτό το ξέρουμε. Και οι τεχνολογίες βελτιώνονται. Όμως θα πρέπει να δούμε τις τεχνολογίες αυτές στο σύνολό τους. Για παράδειγμα, μπαταρίες και συσσωρευτές και αυτοί επηρεάζουν αντικά το περιβάλλον, το βλάπτουν. Οπότε θα πρέπει να γίνει η, μείωση να γίνει ε, οριζοντίως. Ε, πρέπει να μειωθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και από τις μπαταρίες, να μπορούν να ανακυκλωθούν κλπ. Επίσης, να μπορούν να χρησιμοποιούν οι μπαταρίες λιγότερους ε, μολυσματικούς παράγοντες. Θα πρέπει να δώσουμε αυτόν τον τρόπο μια όθηση στις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες για βελτιωμένες απόδοση μπαταρίες και πιο καθαρές μπαταρίες. η αυτοκινητοβιομηχανία με την κατάλληλη έρευνα και καινοτομία θα παράγει αυτοκίνητα, οχήματα τα οποία πραγματικά θα είναι πολύ πιο αποδοτικά και πολύ πιο χρήσιμα. Ε, ευχαριστώ πολύ όλους και όλες τους συνεισηγητές και όλους συγητές. Είχαμε μερικά προβληματάκια, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ και την Κομισιόν που στις δύσκολες στιγμές μας βοήθησε να βρούμε συμβιβασμούς. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ρουμανική Προεδρία που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για την Επιτροπή, η Επίτροπος. Πούλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλωσορίζουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα με τη μαζί σας την έκθεση Γκοζίμπ σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Και εσείς και οι, συνήθειοι και οι σκιώδεις όχι μόνο τώρα, αλλά σε όλη τη διαδικασία, όπως είπατε, η συνεργασία δεν ήταν πάντα εύκολα, ήταν ανοιχτή, με αφοσίωση και με αποτελέσματα. Χάρη στην δέσμευση και την αποφασιστικότητα όλων των τριών εμπλεκόμενων στην νομοθεσία οργάνων είχαμε σωστό, καλό αποτέλεσμα ένα καθαρό πακέτο κινητικότητας. Ο, ο δημόσιος τομέας έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της απομάκρυνσης από τον άνθρακα στις μεταφορές. Η τα λεωφορεία κυρίως, όπου οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 70% της αγοράς. Χρησιμοποιώντας ε, την, ε, τις δημόσιες συμβάσεις για την επιτάχυνση των καθαρών οχημάτων η οδηγία επιτρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για, την μηδενι... για τη συγκινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Κατά την άποψή μα, το κείμενο που συζητήθηκε στον τριμερή διάλογο στι 11 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεύει μια καλή συμβαστική λύση μεταξύ των διαφόρων θέσεων και ε, ετοιμάτων. Δείχνει ότι υπάρχει επαρκή φιλοδοξία αφήνοντα ε, αρκετή ευελιξία για την υλοποίηση ούτω ώστε οι στόχοι της οδηγίας να μπορούν να ελοποιηθούν χωρίς μεγάλο διοικητικό βάρος για τις δημόσιες αρχές. Με την, με την έγκριση της αναθεωρημένης οδηγίας δίνουμε ορισμό ότι είναι καθαρό όχημα και θέτουμε σαφείς στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίω ειδικού στόχους για λεωφορεία μηδενικών εκπομπών. Έχω εμπιστοσύνη στο ότι η συμφωνία που επιτέχθη στον τριμερή διάλογο θέτει επαρκή σαφ, επαρκώς σαφή ορισμό και επαρκώς φιλόδοξους εθνικούς στόχους. Το κείμενο επίσης δίνει μεγάλη ευελιξία για το πώς οι προσπάθειες ε, επιμερίζονται μεταξύ κρατών μελών, επιτρέποντας μία κοστοποτελεσματική εφαρμογή που δεν θα δημιουργήσει σημαντική επιβάρυνση στις αρχές των κρατών μελών. Πολλές πόλεις μας, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, ε, η Βασοβία, το, η Βαρκελόνη, το Μιλάνο, η Λουμπλιάνα, το Μόναχο και πολλές άλλες ήδη έχουν αναλάβει εθελούσες δεσμεύσεις ξεπερνώντας αυτό που απαιτεί η οδηγία. Θα βοηθήσουμε και άλλες πόλεις να ακολουθήσουν το παραδείγμα τους. Η αναθεωρήση θα επεκτείνει και το πεδίο εφαρμογής οδηγίες για να καλύπτονται δημόσιες ε, προμήθειες μέσω πρακτικών όπως ε, ε, ενοικίαση πώληση και σύντομη ενοικίαση. Αυτό θα